Ο Πρόεδρος ε, έθεσε την, ε, το κανονισμό για τα στοιχεία για τις χρηματικές μεταφορές και ύστερα το θέμα του κανονισμού για την ε, χρήση συναλλαγών για ξέπλυμα χρήματος. Και το ισχυει απο από 1η Μαΐου 2015. Καταρχάς έχουμε λοιπόν τώρα την ε, συζήτηση για τη θανατική ποινή στην Ινδονησία. Θα ήθελα